Ξεναρχίζει η συνεδρία. Τα πρακτικά έχουν δυναμηθεί, υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να σχολιάσει. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά.